γίνονται τα πρακτικά αυτά. Η κυρία Ντάμπερ Τεβρούν με ενημέρωσε για την παρέτησή της από τις 3 Μαΐου του 2012 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το σημειώνουμε και σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού του Κοινοβουλίου είναι κενή η θέση της από την ημερομηνία αυτή. Οι αρχές της Ρουμανίας με ενημέρωσαν ότι η κυρία Μνοβάνα Πλούμπ θα αντικατασταθεί από τις 18 Μαΐου από την κυρία Μινόρντα Κλιβέτη. Καλωσορίζουμε λοιπόν αυτήν την νέα συνάδελφο η οποία βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 2 μπορεί να αναλάβει την θέση αυτή. Τα διαπιστευτηριά της δεν έχουν ακόμα εγκριθεί, αλλά βεβαίως ε, θεωρούμε ότι η κυρία Μιναντόρα Κλιβέτη μπορεί να συνεδριάσει